την υποστήριξή του στο website που ανέφερε η κυρία Βορτμαν Κόλλο. Δεν έχω άλλα τέτοια θέματα στην ημερήσια διάταξη, γι' αυτό να περάσουμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη. Η κατάσταση των αστέγων στην Ευρώπη λόγω του κύματο ψύχους. Να δώσω το λόγο εξ ονόματο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λόγο στον Επίτροπο Μπαρνιέ. Κύριε Επίτροπο, έχετε το λόγο. Merci, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι και κύριε συμβουλευτέ, οι συνάδελφοι τη Επιτροπή ε, Μπαρόζο και ο συνάδελφο Άντορ πιο, ε, πιο ιδιαίτερα συμμεριζόμαστε μαζί σα την ανησυχία μα για την κατάσταση των αστέγων στην Ευρώπη λόγω αυτού του κύματο ψύχου. Κανένα δεν μπορεί να μείνει ανέστητο απέναντι στην κατάσταση των όσων κοιμούνται χωρί στέγη κατά τη διάρκεια αυτών των ε, πολύ κρύων νυχτών και ακόμα περισσότερο ε, να μείνει ανάλγητος μπροστά στο θάνατο πολλών ανθρώπων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και γι' αυτό και δικαίως αναρωτιέστε για το τι έχει γίνει για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση και για το τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού απέναντι στις πιο ακραίες αυτές συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Φυσικά, η πρώτη που... Κύριε Επίτροπε, διακόπτει ο Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, με συγχωρείτε, μισό λεπτό παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να φύγετε ησύχως ε, από την αίθουσα και να κάνεις εκτός της αίθουσας. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ κύριε Πίτροπη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Έλεγα λοιπόν ότι όπως το γνωρίζουμε όλοι, η πρώτη, η άμεσα ενδιαφερόμενη για την καταπολέμηση αυτή της, της κατάστασης των αστέγων και που βελτιώνουν την ε, κατάσταση του αποκλεισμού είναι οι αρχές ε, οι τοπικές, όπως εδώ στο Στρασβούργο αλλά και σε άλλα μέρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι αυτές που προσφέρουν ε, ε, επιγόντως καταλήματα. Παντού οι κρατικές και οι τοπικές αρχές κινητοποιούνται. Η κοινή έκθεση του 2010 για την προστασία και την κοινωνική ένταξη καλεί τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν και να συνεχίσουν ε, τα τοπικά περιφερειακά σχέδια ε, για να αντιμετωπίσουν το θέμα των αστέγων και να αντιμετωπίσουν τους ε, τομείς που χρειάζεται να αναλυφθεί δράση γιατί είναι πραγματικά ζωτική σημασία τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια, το γνωρίζουν πολύ καλά και ε, ενεργούν και αντιστοίχω. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό το σώμα αυτό να τονίσει την επίγουσα κατάσταση τοποθετώντας αυτό το θέμα στην μερίσια διάταξη. Αν και οι δυνατότητες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περιορισμένες, έχουμε και εμείς ένα ρόλο να παίξουμε. Καταρχήν να θυμίσουμε στα κράτη-μέλη τις ευθύνες τους και να τα στηρίξουμε στις προσπάθειές τους πιο μακροπρόθεσμα θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα και να βελτιώσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να μετρήσουμε το εύρος του φαινομένου και να ενεργήσουμε έτσι καλύτερα. Για παράδειγμα, μέσω του προγράμματος Progress, η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά στη χρηματοδότηση μιας νέας μελέτης για τη σχέση μεταξύ των Αναστέγων και της μετανάστευσης μέσω της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των ΜΚΟ που εργάζονται με του αστέγους. Η Κομισιόν μέσα στο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο 2014-2020 ε, ζητά και προβλέπει το Κοινωνικό Ταμείο να ανταποκριθεί πιο συγκεκριμένα, πιο στοχευμένα σε αυτό το θέμα των καταλημάτων και της στέγασης των αστέγων. Επίσης ε, προβλέπονται συγκεκριμένα προγράμματα για νέες προσεγγίσεις μέσω εργασιών για την κοινωνική καινοτομία. Ο συνάδελφος Επίτροπος Αντόρ παρουσίασε μια καινοτόμα προσέγγιση που ξεκίνησε μέσω των ε, σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για τη στέγαση ε, ανθρώπων μέσα στους σταθμού. Ε, μέσω ενό κοινού χάρτη οι διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείε έχουν κάνει κοινό πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Ένταξη μέσω της χρηματοδότησης, μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται Ελπίδα μέσα στους σταθμούς και θα συνεχιστεί με ένα πρόγραμμα το οποίο θα αποκαλείται Εργασία μέσα στους σταθμούς. Εμεί χαιρετίζουμε τον χάρτη αυτόν ε, που είναι σε σταθερή αντίθεση με τον αποκλεισμό ε, πρόκειται για μια ευρεία ε, οπτική των κοινωνικών αναγκών που θέλει να λάβει υπόψη την προσθέμενη αξία ε, και τη συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς των ενώσεων και των ΜΚΟ που παίζουν υποδηματικό ρόλο. Οι επιχειρήσει, οι κυβερνήσει, οι τοπικές περιφερειακές αρχές, οι θύνοντες της κοινωνία των πολιτών καθημερινά α φτιάξουμε αυτή την, την κοινωνική Ευρώπη Πράγμα που απαιτείται από την αλληλεγγύη για του ε, αστέγου. Έχουμε ενεργήσει, πρέπει πολλά ακόμα να γίνουν. Η Κομισιόν προσπαθεί να δώσει όσο γίνεται μεγαλύτερη στήριξη από πλευρά τη Ένωση στι προσπάθειε των κρατών μέλων για αυτή την πρόκληση των αστέγων. Βασιζόμαστε κυρίω στι εργασίε ε, του σώματο, όπω εκφράστηκαν στι ε, εργασίε τη 14η Σεπτεμβρίου του παρελθόντος έτους. Επίσης έχουμε δημοσιεύσει Προτάσει τον περασμένο Οκτώβριο με νέα μέσα ώστε οι κοινωνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν καλύτερα να υλοποιήσουν την αποστολή του. και γνωρίζουμε ότι ορισμένε εξ αυτών ασχολούνται με τους άστεγους ε, και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ευάλωτων ανθρώπων όπως είναι οι άστεγοι. Να σα δώσω τρία παραδείγματα καλύτερη χρήση των διευθυντικών ταμείων, απλοποιημένοι κανόνε και λιγότερη έλεγχη για τι κρατικέ ανισχύσει που ε, απευθύνονται στι κοινωνικέ υπηρεσίε που συνοδεύουν τους ευάλωτου ανθρώπου, και έπειτα κανόνε για τους ε, κρατικέ ε, προμήθειε που διευκολύνουν και πάλι του κανονισμού για τι κοινωνικέ υπηρεσίε και ευνοούν τα προγράμματα υπέρ τη ένταξη. Αυτά έχω να σα πω και εξ ονόματο του συναδέλφου Αντόρ και σα ευχαριστώ που επιστήσατε την προσοχή σα σε αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Κυρίες και κύριοι, πρωτού ξεκινήσω τη συζήτηση να κάνω την εξή υπότεξη. Πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο για την διαδικασία Catch the Eye. Θα πρέπει να σας πω ότι στην ημερήσια διάταξη ορίζεται ότι θα γίνει μόνο ένας ε, γύρος ε, ομιλητών των, από εξονόματος των ομάδων. Ε, πολύ λυπάμαι λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαδικασία Catch the Eye. Και τώρα για το ELK... Ο Ιώσεφ Ντόλ, ο πρόεδρος της ομάδας, έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, λέει, εκτός μικροφώνου, ο κύριος Ντόλ. Συνάδελφε Ντόλ, ανάψτε το μικρόφωνο. Για να σα ακούσουμε καλύτερα, να σας καταλάβουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ το εκτιμώ αυτό. Και τώρα, Μιλούμε για περισσότερου από 600 επιθετέ μέρε πέθανε στην Ευρώπη και ήταν και θύματα του ψύχου και κυρίω τη ε, μοναξιά από μόνο δεν είναι ε, επομένω θέμα μόνο οικονομικό, χρηματοπιστωτικό. Η Ευρώπη είναι και υπόθεση αλληλεγγύη. Και επομένω αυτό το κύμα ψύχου το οποίο χτύπησε τον, τον κόσμο μα δίνει την ευκαιρία αυτό να το αποδείξουμε. Και αποδεικνύεται ότι τα αποθέματα τροφίμων τα οποία δίνονται όσον αφορά την επιστηστική αγωγή είναι πάρα πολύ ανεπαρκή και το ίδιο αφορά και τι ενισχύσει για του μη κυβερνητικού οργανισμού αντίστοιχου. Οπότε είμαστε όμοιροι μέχρι το 2013 όμοιροι ενό διεθνού προβλήματο νομική βάση. Επομένω, θα πρέπει να δούμε πώ θα κάνουμε κάτι όσον αφορά αυτό το σκάνδαλο τη διασπάθηση των, των επιστηστικών φόρων. Επομένω. σκεφτείτε στις, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ πόσα, πόσα πετάνε, ενώ υπάρχουν ένα σωρό φορεί που δεν έχουν αρκετά τρόφιμα για να τα διανύμουν. Επομένω, ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι και να θεσπίσουμε αυτό το δίκτυο. Εγώ ήμουν δήμαρχος σε κάποιο χωριό πολλά χρόνια και ξέρω ότι εκεί πέρα παίζεται το παιχνίδι και επομένω χρειάζεται μια, ένα, ένα δίκτυο ε, τέτοια τεχνική βοήθεια όπω το έγινε προσπάθεια τελευταία. Το πιο ό,τι πιο αποτελεσματικό, αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε και πρέπει όμω κάτι να κάνουμε και επίση να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό το πρόγραμμα το επισυντηστικό ε, και επομένω ταυτόχρονα να βοηθήσουμε μια κοινή πολιτική ενέργεια γιατί σήμερα ε, βλέπουμε ότι κόβεται το φυσικό αέριο, κόβεται το ηλεκτρικό για αυτούς που το έχουν ανάγκη, για αυτούς που δεν μπορούν και να το πληρώσουν. Και η αντίδρασή μας ε, σε όλες μας τις χώρες είναι πάρα πολύ βραδία. Επομένως θα πρέπει εκεί να δώσουμε χειραβοηθείας, ε, αγαπητέ Μισελ, να έχουμε αυτό το δίκτυο της ε, προστασίας του πολίτη και το οποίο να είναι και επικαιροποιημένο και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε να μην συζητάμε τα ίδια του χρόνου, μην έχουμε τα ίδια δράματα, τα ίδια κατεπήγοντα. Μια που τώρα γνωρίζουμε τι γίνεται, θα πρέπει στις μη κυβερνού οργανισμού να δώσουμε τα μέσα και επίσης αυτούς τους συμπατριώτες μας που ασχολούνται με το θέμα αυτό και να μην ε, διασπαθίζουμε τους πόρους ε, στους μεγάλους ε, οργανισμούς. Ευχαριστώ κύριε Ντόλ και τώρα από τους σοσιαλδημοκράτες η κυρία Γκυγιώμα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το κύμα ψύχο που χτυπά την Ευρώπη τι τελευταίε εβδομάδε ήδη έχει ε, προκαλέσει πολλά θύματα, κυρίω άστεγου. Και το θέμα αυτό δημιουργεί με πολλά συναισθήματα στην κοινή γνώμη. Γνωρίζουμε ωστόσο πω αποτέλεσαν θύματα αυτή τη επισφάλεια που επικρατεί. Γιατί ναι, το ψύχο σκοτώνει. Όμω πέρα από αυτό έχουμε την κρίση, την φτώχεια και την επισφάλεια που, που σκοτώνει του αποκλεισμένου από την κοινωνία. Τρία εκατομμύρια είναι η μεγάλη περιθεωριακή και άλλο ένα και περισσότεροι ηλικιωμένοι, νέοι, ολόκληρε οικογένειε. Ανάμεσα στου άστεγου βρίσκουμε κάποιες φορές και Σε περίοδο οικονομική κρίση ε, η μετακίνηση προ αυτή την κατάσταση μπορεί να, είναι να γίνει πάρα πολύ γρήγορα για μια οικογένεια που μέχρι τώρα τα έβγαζε πέρα. Έπειτα οι άστεχοι μπορεί να καλύπτουν πολλέ διαφορετικέ πραγματικότητες. Είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται στο αυτοκίνητό του σε ένα ξενοδοχείο που δεν ή που μπορεί ε, προσωρινά να μένουν σε, κάποιο, σε συγγενείς. Αυτό το θέμα καλύπτει ένα ευρύ κοινό και πολλαπλές καταστάσεις. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις γρήγορες και στενάρε. Τι γίνεται, διαβάζω πολύ γρήγορα. Με συγχωρείτε. Υποχρεούμεθα να ενεργήσουμε όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε την επίγουσα ανάγκη, αλλά πιο μακροπρόθεσμα. Αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση, και αυτό είναι ο βασικό μα στόχο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε διευκολύνοντας ανθρώπους να βγουν από τους δρόμους και να δώσουμε καταλήματα στους ανθρώπους που δεν έχουν στέγη. Γιατί διαφορετικά όλοι αυτοί αποκλείονται από διάφορα άλλα δικαιώματα και υπηρεσίες. Η απόγνωσή τους είναι κοινή και η ανάλυση της κατάστασης είναι γνωστή και κοινή. Ας περάσουμε στο επόμενο στάδιο, την πολιτική βούληση. Το Κοινοβούλιο πολλές φορές έχει ζητήσει να σήματιστεί μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική για τους άστεγους Έχουμε την έκθεση του 2010, την έκθεση Μπερές ε, που υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο του 2011 για την ευρωπαϊκή στρατηγική, μια ευρωπαϊκή στρατηγική φιλόδοξη και ολοκληρωμένη. Σκέφτομαι επίση την έκθεση του κυρίου του συναδέλφου Νταρντέν τον περασμένο Νοέμβριο για την φτώχεια και τον αποκλεισμό. Οι ευρωβουλευτέ λοιπόν σα ζήτησαν να φτιάξετε αυτή τη στρατηγική για του άστεγου που θα διαρθρώνεται γύρω από συγκεκριμένου στόχου που δεν θα επαναλάβω τώρα ε, λόγω έλλειψη χρόνου. Πού βρίσκεται αυτό ο δικό χάρτη, πού βρίσκεται, ποια ποσά μπορούν να κινητοποιηθούν από το Κοινωνικό Ταμείο και από το, τα Διαρθωτικά Ταμεία. Ας μην μείνουμε στις ε, δηλώσεις προθέσεων. Δυστυχώ και το 2010 δεν έφερε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα πρέπει η πολιτική του, μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής για το 2020 να συμπεριληφθεί και η καταπολέμηση της επισφάλειας. Δεν μπορούμε να επαφιόμεθα μόνο στην καλή βούληση και στα μέσα των ε, διαφόρων οργανώσεων και ενώσεων. Σε καιρό κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή που επιβάλλει ε, προγράμματα λιτότητα. Δεν θέλουμε βέβαια να πούμε μόνο σε εύκολε λύσει, ότι δίθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μόνο να βοηθήσει και να σώσει τι τράπεζε. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να καταπολεμήσουμε αυτή την καρικοτούρα και να μην ε, ικανοποιηθούμε μόνο με δηλώσει προθέσεων. Είναι ένα θέμα όπου μπορούμε να κάνουμε πολλά και γι' αυτό ζητούμε ακόμα μια φορά μια βολονταριστική δράση και συγκεκριμένη υπέρ των αστέγων. Σας ευχαριστώ. Κυρία δεν χρησιμοποίησατε το χρόνο σας. Μπορούσατε να μιλήσετε πολύ πιο αργά. 30 δευτερόλεπτα νωρίτερα κλείσατε το μικρόφωνο σας. Οι καημένοι διερμηνείς πραγματικά δυσκολεύτηκαν να σας παρακολουθήσουν. Την επόμενη φορά ας μιλήσετε τα τέσσερα λεπτά σας πιο ήρεμα. Ο συνάδελφο Ρινάλδη για τους φιλελεύθερου και δημοκράτες έχει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάπω. Ε, προκλητικά θα μπορούσαμε να ξεκινούσαμε αυτήν την Ολομέλεια με ένα, τηρώντας ενός λεπτού ε, σιγή προς τιμήν των 600 άστεγων που έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα, μέσα σε αυτό το κύμα ψύχου. Σε αυτό το επιφυλάσσουμε μόνο για το διάσημα, τους διάσημους νεκρούς. Ίσως όμως θα είχε υπάρξει μια ένδειξη ευθύνης ε, ε, πολύ συμβολική και πολύ ισχυρή. Δυστυχώ δεν, δεν ξέρω γιατί όλες αυτές οι αξίες τις οποίες εμείς υποστηρίζουμε δεν μπορούν να ισχύσουν για του αστέγου Είτε είναι πολιτε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι. Πολύ συχνά γιατί αυτοί δεν ε, δημιουργούν εκλογικό σώμα και δεν, δημιουργούν, δεν είναι αυτοί στου οποίου οφείλεται η συνένεση. Και επίσης όπω είπε και ο Επίτροπος ε, είναι θέμα των κρατών μελών. Ωστόσο, αποκτά διασυνοριακό χαρακτήρα αυτή η κατάσταση και γίνεται όλο και πιο προφανής. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές επανειλημμένο στην Κομισιόν. Πόσο μπορούν να δοθούν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία συμπεριλαμβανομένων και των Διορθωτικών Ταμείων και του Κοινωνικού Ταμείου για τους αστέγους. Έπειτα, η ελεύθερη κυκλοφορία των αστέγων αυτή είναι πραγματικά εγγυημένη ή είναι δυνατόν κάποιο κράτος μέλος να την περιορίσει ακριβώς γιατί αυτοί οι πολίτες και μιλώ για Ευρωπαίους πολίτες ίσως να μην έχουν σταθερό το ποδιαμονη και έπειτα η μήνυμο βοήθεια και η μήνυμο υπηρεσίες. Κάποια κράτη-μέλη την αρνήθηκαν. Πολίτες άλλων κρατών μελών ε, σε πολίτες μάλλον άλλων κρατών μελών βασιζόμενοι στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Νομίζω, είμαστε βέβαιοι πως αυτό είναι αποδεκτό από νομικής άποψης. Έπειτα η ΦΑΟ όρισε ότι είναι 179 κιλά τα τρόφιμα που σπαταλώνται από κάθε Ευρωπαίο πολίτη ετησίως. Ποια θα μπορούσε να είναι μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να καταπολεμήσουμε αυτή τη σπατάλη. Εγώ πιστεύω πως θα μπορούσε να είναι οικονομική και κοινωνική, αλλά εδώ διακυβεύεται και η ταυτότητα η ευρωπαϊκή. Σας ευχαριστώ κύριε Ρινάλντι. Εξ ονόματος των Πρασίνων έχει τώρα το λόγο η κυρία Καρίμα Μαντέλη για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μπαρνία, αγαπητοί συνάδελφοι, σας το λέω, είμαι οργισμένη. Διότι εδώ και δύο χρόνια έχουμε αυτή τη διάσκεψη τη συνένεση υπό Βελγική Προεδρία ε, χάρη μια στρατηγική για τους αστέους και εδώ στο Ευρωπαϊκό ε, συντάξαμε μια διακήρυξη για τους ε, αστέγους και εγώ έφτιαξα επίσης ένα ψήφισμα για τους αστέγους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας. Ε, όλα αυτά ήσαν νεκρό γράμμα. Και δυστυχώς ε, σήμερα στο Συμβούλιο ε, βλέπουμε άδειε έδρε στο χώρο, στην πτέρυγα τη ολομέλειας με το Συμβούλιο. Τι γίνεται με αυτή την ενίσχυση όσον αφορά τη στέγαση, τι γίνεται με αυτού που δεν έχουν αρκετά χρήματα. Έχουμε αυτό το, το, το κύμα ψύχους και ε, ε, είχαμε 600 που πέθαναν οι περισσότερους. Όμως το θέμα δεν είναι τι θα κάνουμε ε, το χειμώνα, τι θα κάνουμε όλο το χρόνο, τα δικαιώματά τους, τα οποία τα έχουν απεμπολίσει. Λοιπόν, θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε δραστήριοι και αλληλεγγύοι προς τους πιο ευάλωτους. Η κατάσταση δεν είναι απλώς ανησυχητική, είναι πολύ χειρότερα. Στην Ελλάδα 25% ε, σε δύο χρόνια ανέβηκαν οι άστεγοι. Στην Ουγγαρία τους διώκει και τους βάζει πρόστιμα η αστυνομία. Στη Δεγαλία βλέπουμε να θεσπίζονται νόμοι που ποινικοποιούν την ε, ελεημοσύνη, ε, το να ψάχνει κανείς τα φαγιά που είναι πεταμένα στα σκουπίδια. Πού πάμε, βλέπουμε επομένω με αυτές τις πολιτικές λιτότητες των διαφορών κυβερνήσεων ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, αγαπητοί συνάδελφοι ας ε, ε, ε, κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Κύριε Επίτροπε, κάτι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει τον ρόλο που της αρμόζει όσον αφορά την ελεγγύη μεταξύ κρατών και λαών. Επίσης θα πρέπει αμέσω αμέσως να συγκαλέσουμε ένα συμβούλιο των αρμοδίων υπουργών για να σώσουν ανθρώπινες ζωές πριν είναι πολύ αργά. Θα πρέπει να θεσπίσει κάποια μέτρα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα που έχουν το κύμα ψύχους, να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους, τα δε κράτη τα οποία δεν τρούν τις υποχρεώσεις τους για να δώσουν αυτή τη βοήθεια, να τους υποληθούν κυρώσεις. Να μην τους απαγορεύουν το, το να βρουν στέγαση στα άσυλα, μην ποινικοποιούν το, να είναι κανείς άστεγος. Κύριε Μπαρνία, σας το επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει εδώ και τώρα να συγκροτήσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους αστέγους. Είναι σαφής ο στόχος και ο σκοπός, το έχουμε πει και ξαναπεί, κανένας δεν θα πρέπει μέχρι το 2015 να κοιμάται στο δρόμο. Είναι επίγον, κατεπίγον να τους δώσουμε την ευκαιρία να κοιμούνται κάπου. Να σταματήσει αυτή η παγωμένη, παγερή σιωπή των αρμόδιων στην Ευρώπη. Εδώ και τώρα πρέπει να λάβετε δράση. Κόβει το μικρόφωνο ο πρόεδρος. Και τώρα. Για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστάς έχει το λόγο ο κύριος Καρίμ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, τώρα πια όλες οι κοινωνίες και κάθε μία χωριστά κρίνονται από το πώς φέρονται στους πρεσβύτερους και τους πιο ευάλωτους. Έχουμε περίπου Τρία εκατομμύρια αστέγων στην Ευρώπη. Και ακόμα και στον Ευρωβασίλειο τη χώρα μου έχουμε περιπτώσεις υποθερμίας που έχουν πλήξει τους υπέργυρους και έχουν αυτές τις περιπτώσεις διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και είναι επομένω τέτοιος βαθμός προβλήματος που σήμερα δεν με εξέπληξε όταν πήρα μια εφημερίδα μεγάλη κυκλοφορία στο Ρωμαίο Βασίλειο και ο βασικός τίτλος ήταν «Πάγωσε από το κρύο, δεν μπορούσε να πληρώσει τους λογαριασμούς» έχουμε μόνο λοιπόν σε αυτού του αστέγου. Ναι, είναι σοβαρό το πρόβλημα και το δικό μου επιχείρημα είναι ότι άπαξ και θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των αστέχων και εκείνων ε, που γενικά πλήσονται από το κύμα ψύχους θα πρέπει βεβαίως να έχουμε μέτρα και για εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως θα μπορούσαν να καταντήσουν άσταγη μια που όπως είναι τώρα η οικονομική κατάσταση δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Άρα θα πρέπει κάτι να κάνουμε για όλες αυτές τις ε, κατασχέσεις και τις απολύσεις. 233 τελευταίες 7 εβδομάδες είχαμε ε, κάποιους που πέθανε και στη Γαλλία, που είπατε για 600 τελευταίες εβδομάδες. Όλα αυτά θα πρέπει να προξενούν ντροπή. Ο Επίτροπος Μπαγνέ είπε για το πόσο δεν δεμέναν τα χέρια μας στο Υποκοινοβούλιο. Ακριβώς θα πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι με τα κράτη-μέλη, να τους πείσουμε να συντονιστούν για να ακολουθήσουν την καλύτερη, πιο δόκιμη συνταγή. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Και τώρα, για δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Γκαμπρίλε Τσίμερ για την Ευρωπαϊκή Νοτική Αριστερά. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, παρόζω αγαπητέ συνάδελφοι, το ψύχος καταδεικνύει τα κενά στην ε, ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, έχει αποτύχει σε όλες τις γραμμές. Ε, νεκροί πάνω από 600 άνθρωποι στο πολικό ψύχος, 80 νεκροί στην Πολωνία, 130 στην Ουκρανία, εκατοντάδες στη Ρωσία, αλλά και στη Γερμανία βλέπουμε τα πρωταθήματα. Οι πιο πολλοί παγώνουν οι περισσότεροι που πεθαίνουν από το κρύο είναι οι άσταγοι. Παγώνουν ε, κατά γέφυρες, στο δρόμο, σε διαμερίσματα που δεν θερμαίνονται. Δεν μπόρεσαν να πληρώσουν το λογαριασμό του ηλεκτρικού και έτσι τους έχουν κλείσει τη θέρμανση. Όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να, αναλάβουν, να λάβουν κατεπήγοντα μέτρα για να προστατεύσουν όσους είναι ευάλωτοι στο κρύο. Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι δήμικοι κοινότητε για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Και αυτό που θεωρώ ότι είναι το χειρότερο είναι ότι κανείς δεν μπορεί σήμερα να εκτιμήσει ακριβώς πόσοι άστεγοι υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσοι άνθρωποι κινδυνεύουν να παγώσουν από το κρύο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει καμία, κανένας κοινός δείκτης, καμία, κανένα στατιστικό στοιχείο που να μπορεί να καταδείξει πραγματικά τι γίνεται, ούτε καν στη Γερμανία. Ζητούμε να σχηματιστεί task force, ομάδα δράσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταστούν ε, ευδιάκριτες οι ανάγκες όλων των ε, κοινοτήτων. Θέλουμε να υπάρχουν στατιστικοί δείκτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ε, διοργανώνονται γύρω από τις ομάδες που ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προβούν σε ανάλογες νομοθετικές δράσεις. Θέλουμε να επιβληθούν ευρωπαϊκά προγράμματα για την εξυγίανση και την αντιάρθρωση των ε, κατοικιών και προτείνουμε να γίνει συζήτηση για ελάχιστα παραγωγικά πρότυπα και κοινωνικά πρότυπα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπερεύεται κατά πολύ το χρονικό όριο αγόρευση και τώρα πάμε στην τελευταία παρέμβαση. Έχει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει στους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Ο Επίτροπος, κύριος Μπαρνί, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ρενάλντι και άλλοι συναδέλφοι μας είπαν για αυτούς τους 660 οι οποίοι πέθαναν τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορες χώρες και κρίμα που έρχεται κάτι τέτοιο διότι αυτό μας δείχνει το μέγεθος της τραγωδίας τον πανευρωπαϊκό της χαρακτήρα και αυτό σας λέω ότι εκ τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι χρειάζεται επιβάλλεται το Κοινοβούλιο και εμείς να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια απάντηση που αντιστοιχεί στις διαστάσεις του προβλήματος ε, και κυρία όπως γνωρίζετε η βασική μας ε, η βασική αρμοδιότητα μάλλον ε, είναι των κρατών μελών το πρώτο το οποίο απαιτείται σε μια τέτοια προβληματική είναι να λάβουμε το ρόλο μας εσείς και εμείς δηλαδή να πιέσουν τα κρατημέλη τόσο ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όλοι μαζί και το καθένα χωριστά. Επίσης, ο πρόεδρος Ντόλ ανέφερα τη συζήτηση, όπω και ο συνάδελφο Τσόλο, όσον αφορά την εμπιστική βοήθεια. Όμω, τι είναι, γιατί μπλοκαστήκε το πρόγραμμα εμπιστική βοήθεια, το οποίο ακριβώ αφορούσε την ενίσχυση των πλέον βαλόντων και ακριβώ για αυτού του ε, φορεί του οποίου αναφέρατε. Γιατί δεν μιλάω για τίποτα μεγάλα νομικά πρόσωπα. Είναι κάποιοι τοπικοί φορεί που επιτελούν το έργο. Επομένω, τι γίνεται. Είναι κρατική, περιφερειακή η σχετική αρμοδιότητα για την ψυχική βοήθεια. Δεν έχω εμεί αρμοδιότητα, έχουν και όμω ακριβώ λόγω τη δική σα αποφασιστικότητα και λόγω τη δραστηριότητα του συναδέλφου Τσόλο καταφέραμε να πείσουμε περί εκείνου του θέματος το Συμβούλιο. Επομένως, έχουμε αρμόδια κάτι να κάνουμε, κύριε Καρίμ, Ντόλ, σας είπα τι γίνεται για αυτές τις ε, καθολικές υπηρεσίες, τις βασικές, δηλαδή τη στέγαση, την, ε, τον επισητισμό, την κάλυψη ενεργειακών αναγκών. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε με το κανονιστικό πλαίσιο για αυτούς οι οποίοι υποφέρουν και να βοηθήσουμε αυτούς που είναι πιο κοντά στην επιτόπου δράση και όταν ε, είχα παρουσιάσει κάτι που τώρα το στην Κοινοβουλική Επιτροπή όσον αφορά τις ε, κρατικές προμήθειες και τις κρατικές ενισχύσεις ήταν και ο κύριος Σαλμούνια τότε είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπιστεί και ο κοινωνικό αποκλεισμό σε σχέση με αυτέ τι βασικέ καθολικέ κοινωνικέ υπηρεσίε και πώ θα διευκολυνθούν οι υπηρεσίε κοινωνική πρόνοια των κρατών μελών. Να, επομένω, πώ μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει έναν ρόλο. Κυρία Γκυγιόμ, και η κυρία Ντελή μας είπε για κάποια στρατική για τους ε, αστέγους και μας παρακόμψατε και στο ψήφισμα του 2011. Έχω να πω στον κύριο Ρινάλντι ότι από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεσπίζουν κάποια μέτρα. Έχουμε μια μελέτη για την κινητικότητα, τη μετανάστευση, τις κατασχέσεις, στατική για τη στέγαση και επίσης σας είπα το πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τους ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Περιφερειακού Ταμείου ή άλλων ταμείων για την γενική πολιτική. Έχω εδώ πέρα κάποια στοιχεία τα οποία φανερώνουν ότι από το 2007-2013 τα κρατημέλη έχουν δώσει 10 δις από το Κοινωνικό Ταμείο για δράσεις πολέμησης του γενικού αποκλεισμού για τους πιο ευάλωτους της ε, κοινωνίας μας. Επίσης, κυρία Ντελή, συμφωνώ, συμφωνούμε ε, με αυτά τα οποία είπατε για αυτό που γίνεται σε κάποιες χώρες με την ποινικοποίηση, την απαράδεκτη των ε, αστέγων. Και σε κάποια κρατημέλη είχαμε και επιθέσεις κατά αστέγων. Οπότε όπως και εσεί και εμεί θέλουμε να καλούσουμε τα κρατημέλη να λάβουν τις ευθύνε του ενώπιον αυτή τη καταστάσεω. Πρόεδρε Ντόλ λαμβάνει υπόψη. Σημειώνω αυτό που είπε για την ε, πολιτική προστασία. Ξέρετε ότι το θέμα αυτό με απασχολεί ιδιαίτερω. Η κυρία Γεωργίευα έχει αναπτύξει αξιόλογη δράση πάνω σε αυτό και έχουμε διατυπώσει συγκεκριμένε προτάσει, ούτω ώστε κάποια μέρα να μπορέσουμε να υπάρχει αυτό το οποίο οραματίζεστε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και κάποιε θεομηνίε, καταστάσει, καταστροφέ εκτό Ένωση, αλλά και για όσα πλήσουν την ίδια την Ευρώπη και πλήσουν τους πιο ευάλωτους και θα και δεν τον κινδύνο την υγεία, τη δημόσια. επομένω. είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έστω και για λίγο αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία, το συζητήσαμε και έχουμε τα μέσα οικονομικά, πολιτικά, νομικά και γι' αυτό νομίζω ότι μέσα αυτή τη συγκυρία της μεγάλης κρίσης που σοβεί έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι τώρα βρίσκονται στο δρόμο όπως είπε η κυρία μου, και κάποιοι που είναι, γίνονται άνεργοι. Άρα επομένω πρέπει, μπορούμε κάτι να κάνουμε και θα κάνουμε, ότι δεν έχουμε όλες τις αρμονίδες που θα έπρεπε ίσως, να δούμε τι θα κάνουμε με τους πιστικού οργανισμούς, ούτω ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στη σωστή του ευρωπαϊκή διάθεση το πρόβλημα αυτό. Ο πρόεδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Με την παρέμβαση του κυρίου Μπαρνιέ, Ολοκληρώνεται η σχετική συζήτηση και τώρα πάμε στο επόμενο σημείο τις Διατάξεις, Πού είναι η έκθεση του συναδέλφου Μασίπ και αφορά το Γραφείο Εναρμόνισης στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς για